Uh, I think we ought to get started. Uh, can I just announce uh, we've changed the time and we're going to go. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα. Θα ψηφίσουμε τώρα στις 9. Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Απλά ε, ήθελα να σας δω να πανικοβάλλεστε. Τέλος πάντων, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη Οι ψηφοφορίε θα ξεκινήσουν στι 11. Το πρώτο θέμα είναι η έκθεση τη κυρία Φικερέδο για το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και για την προώθηση μια κοινωνία χωρί αποκλεισμού στην Ευρώπη. Σα δίνω λοιπόν το λόγο. Muito obrigada, presidente. Ontem, eh, ontem fizemos ναι. Είχαμε εδώ τον κύριο Επίτροπο και συζητήσαμε μαζί του για θέματα της ε, φτώχειας. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην εργασία μας. Γιατί γεννήουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και πραγματικά είναι αδιανόητο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται ειδικά με το, ναι, με το πρόβλημα αυτό. Πόσο μάλλον εφόσον διαπιστώνουμε ότι οι αριθμοί όλα να αυξάνονται μέρα με τη μέρα και η πραγματικά απελπιστική κατάσταση των φτωχών επιδεινώνεται συνεχώς και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι φτωχαίνουν. Αυτό ισχύει για γυναίκες, παιδιά, και όπως σας είπα όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού τελικά βυθίζονται στην ένδια. Στην έκθεση αυτή την οποία σας παρουσιάζω βασίζομαι στα τελευταία στοιχεία που έχουμε τα στοιχεία της Eurostat τον Ιανουάριο αυτού του έτους τα οποία αναφέρονται στις ε, αποδοχές ε, από το τέλος του 2008. Και βεβαίως ε, αυτή δεν είναι μια ακριβής παρουσίαση της σημερινής κατάστασης. Δεν αντικατοπτρίζεται η τωρινή κατάσταση, γιατί η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η κατάσταση είναι πολύ πιο δεινή από αυτήν που εμφανίζεται στα στοιχεία αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα βασιστώ σε αυτά τα δεδομένα που αντικατοπτρίζουν μεγάλο πρόβλημα. 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, 17% του πληθυσμού της Ευρώπης των 27 χωρών μελών διαβιούν με ένα εισόδημα που βρίσκεται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και ε, η απειλή αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη της ένδυας. Δηλαδή 85 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται. Το 2008 ήταν 85 εκατομμύρια, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα είναι μερικά εκατομμύρια παραπάνω. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε όταν λάβουμε τα στοιχεία για την σημερινή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από το 2000, δηλαδή από τότε που έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία είχε σαν στόχο την προσπάθεια να εξαλειφθεί η φτώχεια. Ωστόσο, πρέπει να διαπιστώσουμε δυστυχώς ότι η ένδια, η φτώχεια, έχει αυξηθεί κατά 2% σήμερα. Είναι μια εξαιρετικά δραματική κατάσταση, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους μέχρι 17 ετών, γιατί τα ποσοστά απειλής της ε, φτώχειας ε, φτάνει στο 20% και σε ορισμένε χώρες όπως είναι η Ρουμανία ανέρχεται στο 33%. Σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία 26%, η Ιταλία και η Λετωνία 25%, στην Ισπανία 24%, στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λιθανία, 23%, στην Πολωνία επίσης 23%, δηλαδή τα χαμηλότερα αποστάγματα στη Σλοβενία, τη Φιλανδία και την Δανία με 2% μόνον φτώχεια. Και όταν μιλούμε για αυτή την ε, κατάσταση, αναφερόμαστε στην ε, κατάσταση μετά την καταβολή των επιδομάτων, γιατί αν δεν το λαμβάναμε υπόψη μας ε, αυτό θα, η κατάσταση θα εμφανιζόταν ακόμα χειρότερη. Και αυτό το διαπιστώνουμε και στην αιτιολογική σκέψη. Δηλαδή πριν από την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων σε νέους ε, των 18 ετών ο κίνδυνος στόχιας είναι 18% και για τους άνδρες 25% και για τις γυναίκες 25%, για τους ενηλίκους δηλαδή. Ε, και οι ηλικιωμένοι εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχεια. Ε, το ποσοστό των ανθρώπων που διαβιούν υπό επισφαλής συνθήκες εργασίας αυξάνεται επίσης ε, δραματικά ή έχουν, έχουν θέσεις εργασίες με χαμηλές αποδοχές. Το 2008 ήταν 8% οι φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το κατόφλι της φτώχειας. Σε ορισμένε χώρες, ωστόσο, αυτά τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα. Στην Πορτογαλία λέει ο Ροστάτ ότι το τέλος του 2008 είχαμε 12%. Και βεβαίως αυτός ο ρυθμός αυτά τα ποστά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αλλά έχουμε και στοιχεία της Αεροστάτ όσον αφορά τις στερήσεις, υλικές στερήσεις. Πρόκειται για τμήματα πληθυσμού που δεν έχουν, για παράδειγμα, θέρμανση στο σπίτι τους ή δεν μπορούν να πάρουν ένα πλήρες γεύμα την ημέρα. Αυτό είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό σε ορισμένες χώρες. Δεν θα αναφέρω όλα αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να βρείτε στην επιλογική έκθεση. Ε, στην αιτιολογική σκέψη ε, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα και τα στοιχεία αυτής της μελέτης πραγματικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι είναι αναγκαίο και κατεπήγον να παρέμβουμε. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν ποικίλα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πρόκειται για μέτρα που όπως σας είπα είναι διαφορετικής φύσης και μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά προγράμματα γιατί η φτώχεια εμφανίζει πολλά πρόσωπα και έχει πολλές πτυχές. Εγώ μίλησα για τα εισοδήματα και μίλησα για τις υλικές ε, στερήσεις. Δηλαδή τώρα έχει κάνει στη διάθεση ορισμένα βασικά ε, πράγματα. Αλλά φτώχεια συνιστά το γεγονό ότι δεν έχει πρόσβαση κανεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, τη δικαιοσύνη κλπ. Δεν πρόκειται δηλαδή μόνο για τα υλικά αγαθά. Φτώχεια σημαίνει να έχει κανεί δυσκολίε, στο να έχει μια πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και όπω σα είπα, το θέμα αυτό έχει πολλέ πτυχές. Η πρόσβαση στο δημοκρατικό σύστημα. Ε, η δυνατότητα να μπορούν να συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι, να ενωθούν ή να συνεταιριστούν. Γιατί υπάρχει ο φόβος και δεν μπορούν έτσι να εκφράσουν τα προβλήματά τους. Και αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες. Η φτώχεια θα πρέπει να θεωρηθεί και να ερμηνευθεί στις ε, διάφορες διαστάσεις της. Αυτό θα ήθελα να το πω εκ των προτέρων όταν μιλούμε τώρα για τις ελάχιστες αποδοχές, το ελάχιστο εισόδημα, αυτό είναι μόνο ένα μέτρο για τις πιο βαριές ε, περιπτώσεις φτώχειας και δεν μπορεί να αποτελέσει μια συνταγή υπανάκια για την επίλυση του προβλήματος της φτώχειας. Θα πρέπει να δούμε το φαινόμενο της ένδυας, της όλες του της αποχρώσεις και διαστάσεις και να προσφύγουμε σε πολλαπλά μέτρα για να το καταπολεμήσουμε. Βέβαια, ένα σημαντικό μέτρο είναι, η εξασφάλιση ε, σωστών συνθήκων εργασία και ο ορισμός ελάχιστων αποδοχών, η εξασφάλιση των συντάξεων, η καταχείριση των συντάξεων για αυτούς που έχουν εργαστεί τους το τέλος της ζωής τους να μπορούν να ζήσουν με μια αξιοπρεπή σύνταξη και να μην διολυστήσουν στην ε, εξαθλίωση και στην ένδια, κάτι το οποίο συμβαίνει με πολλούς συνταξιούχους, για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Επίσης το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ε, καλές υπηρεσίες υγείας, ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Σε ποιο πλαίσιο τώρα τοποθετείτε το ελάχιστο εισόδημα, ελάχιστες αποδοχές Υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες μελέτες που δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα υπάρχει αυτό το όριο των ελάχιστων αποδοχών. Όχι όμως, δεν ισχύει όμως σε όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες που δεν... Ε, υπάρχουν ορισμένε χώρες που έχουν λάβει αυτά τα ε, μέτρα και τα αξιοποιούν για την καταπολέμηση της φτώχειας και υπάρχουν σχετικές μελέτες που δείχνουν ότι αν, όταν δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτή η εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου αποδοχών αυξάνεται, διονγκούται το φαινόμενο της φτώχειας. Γι' αυτό είναι σημαντικό όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσουν, να προβλέψουν ένα όριο των αποδοχών, ούτως ώστε οι πολίτες τους να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο καλούμεθα να συζητήσουμε εδώ. Δεν μπορούσα να σας παρουσιάσω περισσότερες προτάσεις σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν κάποια όρια και ε, θα τα δούμε σε αυτή την έκθεση. Αλλά με τις εισφορές των συναδέλφων και μέσω και της δικής μου συμβολής ε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, να εμπλουτίσουμε την έκθεση με πολύ περισσότερα στοιχεία. Αλλά βεβαίως δεν μπόρεσα να το κάνω σε αυτή την πρώτη φάση και ήταν αναγκαίο βεβαίως να πετύχουμε και μία συνένεση ούτε ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να μπορεί να υποστηριχθεί από το σύνολο της Ευρωβουλής. Θα ήθελα να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό υπάρχει εδώ αρκετό περιθώριο επίτευξης μια συνένεσης. Δεν ήθελα να περιοριστώ στην παρουσίαση ενός ε, συγκεκριμένου εργαλείου αλλά το ενδιαφέρον μου στρέφεται σε μια πιο πλατιά προσέγγιση αυτού του θέματος. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι βεβαίως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και μπορούμε να δώσουμε και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρω ότι το επιθυμούν πολλοί συνάδελφοι και υπάρχει και σχετική πολιτική βούληση αλλά τώρα έχουμε μια καλή βάση για να το κάνουμε. Είμαι πολύ προσπεπισμένη ότι σε μια μεταγενέστερη φάση θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ε, προτάσεις και ενδεχομένως θα καταλήξουμε σε μια πλατιά συνένεση για να υποστηριχθεί η έκθεση αυτή κατά τη διάρκεια αυτού του έτους πολέμηση της φτώχειας, ούτως ώστε να αποτελέσει μια σημαντική καθοριστική συμβουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Uh, thanks very much, Mrs. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιγκερέιδο. Βρίσκω εξαιρετική την έκθεσή σας. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μου. Ε, το πρώτο σημείο είναι η παράγραφος F, πολύ, σιγματάφ. Πολύ σωστά λέτε ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν από την ε, φτώχεια, την ένδια. Ε, θα ήθελα όμως να συμπεριλάβω και άλλες ομάδες, ε, τους ηλικιωμένους για παράδειγμα, που επηρεάζονται δυσανάλογα και πολύ συχνά υποφέρουν εξίσου με τις γυναίκες δυσανάλογα δηλαδή με άλλους τομείς του πληθυσμού. Επίσης, ε, μου αρέσει η παράγραφος 5 όπου ζητάμε να ξεκινήσει κάποια πρωτοβουλία ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν κάποια προγράμματα εισοδηματικά για να καταπολεμήσουν την ε, ένδια. Έχω και εγώ κάποιες ιδέες. Ξέρω ότι μιλήσατε λίγο για το θέμα αυτό. Αν μπορείτε όμως να γίνετε πιο συγκεκριμένοι όταν συνοψίσετε αφού ακούσουμε ε, τις παρατηρήσεις όλων των άλλων. Ε, παράγραφος 7 ε, διασαφηνίζει το πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται από την φτώχεια να συμμετέχουν στη διαδικασία λήξης αποφάσεων. Ε, είναι σημαντικό όταν μιλάμε για, την, ε, για τους φτωχούς, για τους άστεγους. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια διάσκεψη για τους άστεγους. Και είδαμε ότι οι άστεγοι αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το πώ δηλαδή εκείνοι θεωρούν ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα μπορέσουν να του βοηθήσουν. Είναι λοιπόν σημαντικό οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τα προβλήματα τη στόχια είναι σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν σχετικοί φορεί, ε, υπάρχουν ε, Υπάρχουν κάποιοι γενικοί φορεί, υπάρχουν όμω και μεμονωμένοι ε, οργανισμοί, φορεί που θέλουν ε, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήξη αποφάσεων. Έχω ήδη ε, συνομιλήσει μαζί του. Χαίρομαι πολύ για το πώ έχει έκθεση αυτή τη στιγμή. Θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε. Αλλά ειλικρινά σα το λέω, βρίσκω εξαιρετική την έκθεση αυτή. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα... Ήθελα να ακούσω τι απόψει σα, ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία των κρατών μελών ε, όσον αφορά το, ε, τα εισοδήματα. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Γκρίνη. Μάλιστα κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με αυτό το σημαντικό θέμα γιατί είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους ε, να τους παραγκονίσουμε σε μια, στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών. Όσον αφορά τώρα τις ελάχιστες περιγράψω την γαλλική εμπειρία όπου προβλέπονται αυτές οι ελάχιστες αποδοχές για την ένταξη των εργαζομένων. Δυστυχώς, στο πλαίσιο αυτό παραμελήθηκε η διάσταση της επανεισδοχής στο χώρο εργασίας. Και τελικά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι οι άνθρωποι τελικά βασίστηκαν ε, σε αυτές τις ελάχιστες αποδοχές που βεβαίως είναι αρκετά ισχνές. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όλο αυτό να περάσει και από μια κοινωνική αναγνώριση και μια εξασφάλιση θέση εργασία. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίε όσον αφορά την επάνωδο στην αγορά εργασία. Η κυρία Πρόεδρος αναφέρθηκε σε άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκες. Ε, θα πρέπει και τα άτομα αυτά να έχουν ε, επαρκή κοινωνική βοήθεια για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και κυρίως να ξαναγυρίσουν το χώρο εργασίας. Αυτό περνά βεβαίω από την ε, κατάρτιση, όχι από μια οποιασδήποτε, ή συγγνώμη, κατάρτιση, γιατί πολύ συχνά αφήνουμε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν ε, διάφορες ε, να κάνουν κάποια κατάρτιση, η οποία τελικά όμως δεν καταλήγει στην αγορά εργασία και δεν του εξασφαλίζει μια θέση εργασία. Θα πρέπει η κατάρτιση αυτή να είναι σε συνάρτηση με, τα, τη, νέα, με τη ζήτηση που υπάρχει για τις νέες θέσει εργασία. Επίσης, ε, για τις συντάξεις θα πρέπει να σκεφτούμε. Άνθρωποι που, έζησαν, που εργάστηκαν όλη τη ζωή και τελικά έχουν ανεπαρκείς συντάξεις, θεωρώ ότι το φαινόμενο αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν επίση στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα πρέπει λοιπόν να τους ξεχνάμε. Τέλος, η φτωχή μισθωτή, γιατί εγώ γνωρίζω καταστάσεις όπου... Ε, άνθρωποι ε, που ζουν από κοινωνικά επιδόματα τελικά βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ανθρώπους που εργάζονται αλλά έχουν ελάχιστες αποδοχές, δηλαδή αποδοχές που τους εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή και υπάρχει αυτό το χάσμα. Τέλος, στην ανάλυση της στόχης που μπορούμε να κάνουμε, ε, συχνά έχουμε το φαινόμενο υπερχρέωσης με ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε ένα αδιάξοδο και θα πρέπει να σκεφτούμε αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δανείζουν χρήματα χωρίς να λάβουν υπόψη την δυνατότητα επιστροφής αποπληρωμής αυτών των δανείων. Και τελικά έρχονται να τους ζητήσουν αυτά τα χρήματα και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν δανειστεί χρήματα δεν έχουν πλέον τα ελάχιστα για να ζήσουν. Θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το φαινόμενο της υπερχρέωσης που είναι ένα πραγματικό αίτιο φτώχειας της κοινωνίας μας. Ε, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και βεβαίως θα συμμετάσχω με δικές μου τροπολογίες στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Jean Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Συμφωνώ με κάποιες παρατηρήσεις που ήδη έγιναν. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Πρόκειται για ρόλο που υποτίθεται ότι έχουν τα εθνικά σχέδια δράσης. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον η Επιτροπή μας να εξετάσει σε τι βαθμό τα εθνικά μέτρα δράσης ε, φροντίζουν για την συμμετοχή των ανθρώπων που ε, ζουν ε, στην Ένδια ή που επηρεάζονται με άλλο τρόπο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Θα ήθελα να πω και κάποια άλλα πράγματα για την έκθεση αυτή, διότι νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποια όπου ακόμα και αν εξετάσουμε τα επίπεδα των επιδομάτων όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, της συντάξης, ε, της ε, παροχές προς άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολύ συχνά ε, τα επίπεδα αυτά βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς τα κράτη-μέλη καθορίζουν τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και ποιες είναι, ποιοι είναι οι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Ήλτα εδώ για το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει δηλαδή στην καταπολέμηση της στόχιας να ε, φροντίσουμε να μην διατηρούμε ανθρώπους σε τέτοια επίπεδα φτώχειας δηλαδή. Ε, επίσης ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε το χάσμα των εισοδημάτων, την ψαλίδα των εισοδημάτων διότι φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό παράγοντα από ό,τι έχουν δείξει μελέτε όσον αφορά την κοινωνική συνοχή και την κοινωνία στο σύνολό τη. Θα ήταν χρήσιμο ίσως να το εξετάσουμε αυτό περαιτέρω. Και ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια ε, νωρίτερα ε, είναι ε, κάποιες περικοπές επιδομάτων στις οποίες βασίζονται πολλοί οι άνθρωποι. Όσον αφορά το πέρασμα από τα επιδόματα στην απασχόληση. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε δηλαδή τα επιδόματα να, ε, να μην αποτελούν εμπόδια την απασχόληση, αλλά δεν είμαι βεβαία εάν αυτό ανήκει πράγματι στην έκθεση αυτή. Είναι πάντως ένα θέμα το οποίο έχει εξετάσει στο παρελθόν η Επιτροπή μας. Πάντως, ε, ενώ στηρίζω τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται. Θα με ενδιαφέρει και η δυνατότητα μιας οδηγία πλαίσιο για τα, ε, για τα ελάχιστα εισοδήματα και θα με ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι πιο, πιο συγκεκριμένο από απλά μια έκκληση να ληφθούν μέτρα. Θα με ενδιαφέρει να δω αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αυτό το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοπεράτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι εισηγητές... Συγγνώμη, η δουλειά της εισηγήτριας είναι εξαιρετική και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. είναι το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε ένα ευρύ αναλυτικό πλαίσιο. Με επιχειρήματα τα οποία να υποστηρίζονται από δεδομένα. Όπως είπε η συγγήτρια, θα μπορούσαμε το πλαίσιο αυτό να το διευρύνουμε περαιτέρω. Νομίζω πάντως ότι η, η συγκήτρια έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Χρήσιμο θα ήταν για όλους μας να προσπαθήσουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αν είναι δυνατόν αναλυτικές προτάσεις, διότι βλέπουμε από τα δεδομένα που έχουμε ότι η φτώχεια είναι ένα πολύ ευρύ φαινόμενο και πολύπτυχο. Δεν μπορεί ένα μέσο να λύσει το πρόβλημα ή να περιορίσει το, τα αποτελέσματα της φτώχειας. Χρειαζόμαστε μια σειρά εργαλείων και κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να συνδέεται με μια συγκεκριμένη κατάσταση. ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα το θέμα. Στον πίνακα της κυρίας Φικερέιδο φαίνεται σαφώς ότι όσον αφορά την ηλικία, τα βασικά προβλήματα επηρεάζουν από τη μία μεριά τα παιδιά και τους εφήβους και από την άλλη τους ε, ηλικιωμένους. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο για τις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες. Θα πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις. Νομίζω ότι το σημαντικότερο για τους νέους είναι η οικογένεια. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, θα πρέπει να εξετάσουμε τις κοινωνικές πολιτικές. Και αυτό που συνενώνει αυτά τα δύο άκρα του φάσματος και αυτό που βρίσκω εγώ πολύ σημαντικό είναι ο ελάχιστος μισθός. Υπάρχουν ε, στα διάφορα κράτη-μέλη διαφορετικές ρυθμίσεις για το θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσε η εισηγήτρια να παρουσιάσει έναν πίνακα που να δείχνει τις διαφορές ανάμεσα στη ρύθμιση στα διάφορα Και θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στα μέτρα υποστήριξης της οικογένειας και τα μέτρα υποστήριξης των ηλικιωμένων. Όπως είπε η κυρία Γκρούνη, είναι διαφορετικά τα μέτρα. Ε, ο κόσμος στην Ευρώπη εργάζεται, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει το κατόφλι της στόχιας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ε, στην Ήπειρό μας. Ε, μιλούσαμε για εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στον ελάχιστο μισθό διότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συστήματα και το κόστος μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με τις προτάσεις της Κομισιόν. Γι' αυτό οι προτάσεις που θα υποβάλουμε θα πρέπει να συνοδεύονται και από μακροοικονομικούς υπολογισμούς. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι η κοινωνική συνοχή ε, σημαίνει οι αποκλεισμένοι να ενταχθούν στην κοινωνία. Στην Ήπειρό μας δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα και δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέρος του πληθυσμού μας που να ζει στην φτώχεια. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό, ε, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές ε, ιδεολογίες στα διαφορετικά μέλη, αλλά είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό που θα πρέπει να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I also... Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Really we... Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για σημαντική έκθεση και η οποία συνδέεται στενά με τη στρατηγική του 2020 το επόμενο εξάμεινο θα χρειαστούμε και πολύ ισχυρή βελγική προεδρία διότι η προτεραιότητά της ε, είπε ότι είναι απόφαση του Συμβουλίου για το ελάχιστο εισόδημα. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να επιδιώξει και η επόμενη Προεδρία ε, τον ίδιο στόχο. Δεν μπορούμε όμως βέβαια να την επηρεάσουμε. Σημαντικό ερώτημα είναι η σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τον καθορισμό του των δικτών ε, του ελάχιστου εισοδήματος. Ε, αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε την ε, διαφορά ανάμεσα στο ελάχιστο εισόδημα και στους ελάχιστους ε, μισθούς. Θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό αποτελούν κίνητρο οι παράγοντες αυτοί κατά την επιλογή εργασίας, διότι νομίζω ότι σε κάποιες χώρες είναι πολύ μικρό το χάσμα είναι πολύ μικρή η διαφορά. Ε, χρήσιμο θα ήταν να έχουμε σχετική επισκόπηση για τα επιμέρους θέματα. Δεν θα ανέφερα εγώ συγκεκριμένες χώρες. Αν έχουμε πίνακα που δείχνει τις διαφορές, νομίζω θα έχουμε συνολική εικόνα. Ε, το να επιλέγουμε κάποιες χώρες μόνο είναι κάπως ε, λεπτό θέμα, είναι κάπως προβληματικό όσον αφορά το σημείο ε, Ζ. Μιλάμε για ομάδες ε, μειονεκτικές, ε, μετανάστες κλπ. Και όσον αφορά την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης υψηλού εισοδήματος, ποια είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να ε, ε, έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας οι άνθρωποι. Και όσον αφορά την πολιτική συνοχή, ε, πώς να αντιμετωπίσουμε τις εδαφικές διαφορές. Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε περισσότερο την σχέση ανάμεσα στην φτώχεια και στις διακρίσεις. Ε, σε πολλές χώρες, στις περισσότερες νομίζω, τα δύο αυτά πράγματα συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την έκθεση αυτή προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Εισήγητρια, και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη των συναδέλφων που εξέφρασαν ε, λέγοντας ότι, ότι η έκθεση αυτή συνιστά μια καλή βάση εργασίας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Και βεβαίως δεν θα ήθελα να επαναλάβω διάφορα πράγματα τα οποία ήδη υπόθηκαν από τους συναδέλφου της δικής μου ομάδας. Παρ' όλα αυτά θα υποσημάνω δύο-τρία στοιχεία. Καταρχήν θεωρώ ότι η έκθεση αυτή μας επιτρέπει να προωθήσουμε στο επίπεδο της ε, αρχαιολογικής έκθεσης τον τεράστιο κίνδυνο της φτώχειας, συγκεκριμένα όσον αφορά ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, κάτι το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με τους νέους, τους ηλικιωμένους κλπ, καθώς και την ε, σημασία να ε, τους εξαφολίσουμε μια πρόσβαση στην αγορά εργασία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλειας, για το συνολικό σύστημα και την κοινωνική ισορροπία. Επίσης αναφέρατε την ε, φτώχεια των γυναικών, τους κινδύνους εδώ, καθώς και στο επίπεδο ορισμένων πιο ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού, κάτι που αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία ορισμένων στοιχείων που υπογραμμίζεται στην αιτιολογική σας έκθεση, όπως είναι ο ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, των ποιοτικών δημοσίων υπηρεσίες, της εξασφάλισης μιας αξιοπρεπούς απασχόλησης, μια σειρά στοιχείων στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε όταν ομιλούμε για τη φτώχεια και επίσης την διάσταση της πολιτικής προτεραιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο Πολιτική προτεραιότητας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στα στοιχεία αυτά. Τώρα, όσον αφορά τι υποδείξει σχετικά με την ίδια την έκθεση, θα ήθελα να πω τα εξή. Euh, όταν αναφέραμε τις, ε, όταν αναφέραμε τους στόχους που, θέλ, που θέλουμε να επιτευχθούν για τη μείωση της φτώχειας, και αναφέρεστε στη συγκεκριμένη στρατηγική 2020 και το διπλασιασμό των 20 εκατομμυρίων σε 40 εκατομμυρία. Ελπίζω ότι θα διατηρηθεί ο στόχος αυτός όσον αφορά τους αριθμούς, αλλά θα πρέπει να δούμε επίσης και τις αναλογίες, τι γίνεται με τις αναλογίες, ώστε στις διάφορες χώρες να υπάρξουν κάποιοι επιτεύξιμοι στόχοι πέρα του συνολικού, του κοινού στόχου. Τα 40 εκατομμύρια είναι πολύ καλός στόχος. Άλλο θέμα, άλλο στοιχείο, όταν αναφέρεστε σε πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Νομίζω εδώ θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε περισσότερο αυτές τις παραγράφους και να επιμείνουμε ούτως ώστε να είναι οι δυνατόν δεσμευτικές πρωτοβουλίες για τις χώρες. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό. Τέλος θα έλεγα ότι συνολικά η έκθεση αυτή προβάλλει πολύ σωστά το ρόλο και την σημασία του επίπεδου ελάχιστων αποδοχών για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση ορίζοντας ένα θεμελιώδη άξονα των ελάχιστων αποδοχών στο πλαίσιο της πάλης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και ε, θεωρώ ότι αυτό δεν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ε, σε αυτή την πρώτη διατύπωση της έκθεσής της. Ίσως θα μπορούσαμε μέσω των τροπολογιών να ενισχύσουμε αυτό το αίτημα της εξασφάλισης ενός επίπεδου ελάχιστων αποδοχών. Βεβαίως, ε, περιτέβει να πω ότι βρίσκομαι στη διάθεσή σας για την, ε, εκπόνηση αυτών των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ε, ε, ο κύριος Χάντλ. Η συνάδελφος Κρούνη και η συνάδελφος Λαμπέρ είπαν ότι στην συζήτηση αυτή βασικό θέμα είναι το πώς οι άνθρωποι μπορούν να απελευθερωθούν μόνοι τους από την φτώχεια. Υπάρχουν πράγματι κατόφλια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους να διατηρήσουν το κοινωνικό τους επίδομα αντί να αρχίσουν να εργάζονται. Θα ήταν λάθος εάν ακολουθούσαμε την κατεύθυνση που συχνά βλέπουμε στον τύπο με μεγάλο γράμματα ότι ε, είναι πολύ ψηλά δηλαδή τα κοινωνικά επιδόματα. Νομίζω ότι ε, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξής. Τα κοινωνικά επιδόματα δεν είναι υπερβολικά υψηλά, αλλά υπάρχει ένα επίπεδο μισθών σε όλα τα κράτη-μέλη που έχει πέσει τόσο χαμηλά που δεν αξίζει τον κόπο για τους ανθρώπους να αρχίσουν να εργάζονται. Οι εργοδότες δηλαδή ε, πληρώνουν μισθούς από τους οποίους δεν μπορεί να ζήσει κανείς και γι' αυτό το θέμα του ελάχιστου μισθού που ανέφερε ο συνάδελφος Γκένσερ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερος παράγοντας που είναι επίσης σημαντικός είναι ότι υπάρχουν νέες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι Δεν αξίζει τον κόπο να εργάζεται κανείς επειδή το φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος ε, είναι τόσο μεγάλο που τελικά καταλήγουν να βγάζουν λιγότερα χρήματα από ότι ε, αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για παράδειγμα από το κράτος ή, άλλες, ε, ή άλλα τέτοια επιδόματα. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα του βασικού μισθού, του ελάχιστου μισθού είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν το κατόφι της στόχιας. Θα πρέπει να προσαρμόσουν επίσης ε, τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές ώστε να αξίζει τον κόπο για τον κόσμο να εργάζεται. Δεν θα πρέπει όμως να γελιόμαστε γενικά για τους ανθρώπους που, ζητούν, που αναζητούν εργασία ή που είναι άνεργοι στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ λίγες θέσεις απασχόλησης ε, και γι' αυτό το ελάχιστο εισόδημα και όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα θα πρέπει να είναι μόνο ένα μέτρο. Ε, υπάρχουν και τα θέματα της πολιτικής που αφορά την, ε, ε τις ώρες εργασίας. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα μέτρα για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πριν... Ε, να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Φιγκερέιδο να, να ρωτήσουμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Κέβιν Ντέντ. Έγιναν κάποιε προκαταρκτικέ μελέτε σχετικά με την φτώχεια σε σχέση με την παρούσα οικονομική κρίση. Η Κομισιόν ε, θα παρουσιάσει μελέτε. Um, um, Η Κομισιόν, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, παρακολουθεί τα αποτελέσματα της κρίσης, τον αντίκτυπο της κρίσης στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα της φτώχειας ε, και του κινδύνου της στόχιας. Ε, όπως εξήγησε ο Επίτροπος χθε, υπάρχουν περαιτέρω πρωτοβουλίε για να προωθηθεί η δουλειά στον τομέα αυτό, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο σωστή και στενή παρακολούθηση του θέματος. Οι δουλειέ αυτές συνεχίζονται. Οι καρποί τη δουλειά αυτής ε, έχουν εν μέρη δημοσιοποιηθεί, άλλοι θα δημοσιοποιηθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέιδο. Ehm, ehm, ναι, όσον αφορά τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε και νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή θα ακούσουμε πολλές προτάσεις στον να που Τώρα, ε, στην αιτιολογική έκθεση όσον αφορά το φαινόμενο της φτώχειας σκέφτηκα ποιες απαντήσεις είναι δυνατόν ε, να δοθούν αλλά δεν είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να τις αναπτύξω. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν εδώ. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να καταπολεμήσει το φαινόμενο της φτώχειας εκείνων που εργάζονται και παρόλα αυτά παραμένουν φτωχοί. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να επεκτείνεται διαρκώς. Βεβαίως χρειαζόμαστε ποιοτικά υψηλή εργασία που να οδηγεί στην εξασφάλιση ορισμένων δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους και όπως υπόθηκε χρειαζόμαστε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ε, αυτό βεβαίως το φαινόμενο εκφράζεται διαφορετικά στην κάθε χώρα αλλά θα πρέπει να είναι μια ποιοτική εργασία που να οδηγεί στην κατοχήρωση ορισμένων δικαιωμάτων. Για να, παράδειγμα, τι γίνεται στη δική μου χώρα. Δεν ε, αρκεί να έχουμε ένα ελάχιστο ύψος αποδοχών. Και όπως σας είπα, αυτό ισχύει για το 12% του πληθυσμού. Βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε ένα κατώτατο όριο αποδοχών, ιδιαιτέρως για γυναίκες που ε, εργάζονται και παίρνουν αυτές τις αποδοχές. Δηλαδή, ε, θέσει εργασία υψηλή υψηλής ποιότητας που να κατοχυρώνουν δικαιώματα για του εργαζόμενου Όταν κάνω αυτή τη διατύπωση αυτό ακριβώ εννοώ. Μια άλλη κατηγορία είναι οι νέοι οι οποίοι δεν θα πρέπει να δουλεύουν, να κάνουν πρακτική εξάσκηση τρεις μήνες, έξι μήνες ή ένα ή δύο χρόνια χωρίς απολύτως καμία αποζημίωση. Καμιά φορά ε, τους δίνουν ένα γεύμα ή δωρεάν εισιτήρια στα μεταφορικά μέσα. Αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για πολλά χρόνια χωρίς απολύτως καμία αμοιβή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Όπως σας είπα, υπάρχει μια έκθεση για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ Επίσης, η μερική εργασία που δεν είναι επιθυμητή από τους εργαζόμενους που τελικά συμπληρώνεται με τα επιδόματα. Φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται, οι λεγόμενες επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Και εδώ θα πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις. Εγώ δεν μπορούσα να τα περιγράψω όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να το συμπληρώσω, να συμπληρώσω την έκθεσή μου, τονίζοντας αυτό το θέμα. Ίσως μπορείτε να το κάνετε εσείς μέσα των τροπολογιών. Οι, οι συντάξει. Οι συνταξιούχοι επίσης θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένο ένα ελάχιστο ύψος αποδοχών ε, συντάξεων για να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς και μετά τη συνταξιοδότησή του. Και αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα. Αλλά δεν είχα το χρόνο για να καλύψω όλα αυτά τα θέματα, αλλά θα το κάνω μελλοντικά. Ή το θέμα που έθεσε ο κ. Γκομφεράτη, το ζήτημα του κόστους. Με αυτό θα ασχοληθώ στο τέλος. Και μετά άλλα, τα άλλα θέματα, οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες, αναφέρονται κάπως γενικόλογα, αλλά δεν δίδονται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους που σας προανέφερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους ανέργους και θα πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές παροχές. Μια αξιοπρεπής εργασία θα πρέπει να αποτελεί ένα κίνητρο Ε, Βεβαίω όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ε, μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασία, οι χρόνια άρρωστοι, οι άνθρωποι με αναπηρίε. Γι' αυτού θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα. Και θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα απασχόληση για του ανθρώπου με αναπηρίε και ε, αξιοπρεπείς αποδοχές για να μπορούν να ζήσουν. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση Υπάρχουν διάφορε δυνατότητε εξασφάλιση των ελάχιστων αποδοχών. Το είπαμε αυτό. Ε, τώρα, τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε ένα ελάχιστο όριο αποδοχών. Ε, ίσως το ποσό δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε το ίδιο γιατί υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Αλλά θα πρέπει αναλογικά να είναι το ίδιο ποσοστό, δηλαδή ένα ποσοστό του ΑΕΠ να οριστεί. Θα ήθελα να αναφέρω, να θέσω εδώ αυτό το θέμα, γιατί σίγουρα θα συζητηθεί πολύ στο μέλλον. Επίσης μιλήσατε για το θέμα του κόστους. Πώς μπορούμε να το εγγυθούμε για χώρες που ήδη είναι πολύ χρεωμένες. Πώς μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος όλα αυτά σχετίζονται με την ε, κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ευρωπαϊκή ελληνική και θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα ε, να ληφθούν τα χρήματα αυτά από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα καινούργια, αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά να πετύχουμε μια συνένεση. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να παίξουμε το ρόλο που πρέπει. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια σχετική διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, θα ακολουθήσει η συζήτηση και θα δούμε. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να πάει τόσο μακριά. Δεν support ε, princípios ε, na minha opinião, deviam ser estes que eu acabo Επίσης, θα πρέπει να, εφόσον υποστηρίζουμε μάλλον αυτές τις αρχές, μπορούμε να πάμε παραπέρα. Γιατί αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης Φτώχειας ε, δεν θα, δεν θα φέρει αποτελέσματα. και ούτε σε 10 χρόνια δεν θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Αντίθετα θα διονγκούται συνεχώς το φαινόμενο αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε μια ξεκάθαρη απόφαση και εδώ ελπίζω να έχω την υποστήριξη των συναδέλφων ούτως ώστε να προχωρήσουμε ώστε το δυνατόν μακρύτερα με τις προτάσεις μας. Γιατί δεν είναι αρκετό το να μας λέει η Επιτροπή ότι ένα χρόνο μετά την κρίση ακόμα βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις. Αλλά τα τελευταία δεδομένα που έχουμε είναι από το 2008, όπως σας είπα. δυστυχώ, δεν έχουμε άλλα στοιχεία στη διάθεσή μας. Οι έρευνες για την αξιολόγηση της φτώχειας είναι ακόμα παλαιότερες. Είναι δεδομένα του 2007. Όλα αυτά δεν ε, σχετίζονται καθόλου πλέον με τη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να σας ε, συστήσω με να προσδώσουμε μια κατεπίγουσα μορφή στις έρευνες για την μελέτη της φτώχειας στις χώρες μας. Σε ορισμένες χώρες η κατάσταση είναι εξαιρετικά δεινή. Γι' αυτό αναφέρομαι σε μέτρα αλληλεγγύης. Και σας παρουσίασα ποιες είναι οι ιδέες μου. Ε, προτάσεις που δεν τις έχω αναπτύξει εδώ. Αλλά περιμένω και τη δική σας συμβολή, ούτε ώστε να προχωρήσουμε όλοι από κοινού. Πολύ. Ε, στις 5 Μαΐου είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Η συζήτηση για τις τροπολογίες την 1η Ιουνίου ε, η έγκριση στις 24 Ιουνίου και ε, νομίζω ότι στις 17 Οκτωβρίου που είναι η μέρα για την εξάλληψη της φτώχειας θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του Όλε Κρίστενσεν για, τις, ε, για την πολιτική αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την τελευταία φορά στην Επιτροπή μας ε, υιοθετήσαμε γνωμοδότηση για το κομμάτι ε, της οδηγίας περί ε, κεφαλαιακών απαιτήσεων που έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό τομέα και κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνέχεια στην γνωμοδότησή μας. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά καλά πράγματα στην έκθεση της Επιτροπής ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ο εισηγητής Ελ Καντράουι έχει συμπεριλάβει θέματα τα οποία επανειλημμένα έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Απασχόλησης. Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι γνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας ε, μιας ανεξάρτητης επιτροπής ε, αμοιβών και επίσης αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που θα εποπτεύει και σε συνοριακό επίπεδο ώστε ε, που θα υποπτεύει αυτό το σύστημα ε, κινδύνου. Παρότι υπάρχουν καλά στοιχεία στην ε, έκθεση, πιστεύω ότι μπορούμε να ε, βελτιώσουμε λίγο τη διατύπωση σε κάποια σημεία. Ε, όπως είπαμε, παλαιότερα στην Επιτροπή Απασχόλησης θέλαμε οι οψιών για τις μετοχές να καταργηθούν τελείως. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων δεν τόλμησε να προχωρήσει μέχρι εκεί, αλλά και σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο ε, επιχειρήσεις και ε, στον ε, και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα διότι οι οψιόν στις μετοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου και προτείνω να καταργηθούν τελείως στις μεταβλητές αμοιβές, στις μεταβλητές αποτοχές. Ε, διότι έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που ε, επιφέρουν ε, αυτά τα μέσα και τα άλλα παρόμοια συστήματα. Φυσικά δεν μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα συστήματα μπόνους, ούτε πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Το α και το ω όμως είναι οι επιπλέον αποδοχές να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη προσπάθεια και γι' αυτό σημαντικό είναι να έχουμε αυτά τα μέσα το clawback ώστε ενδεχομένως να πρέπει κανείς να επιστρέψει χρήματα ε, και όπως είπαμε ε, θέλουμε αυτά να υπολογίζονται μακροπρόθεσμα. Έχουμε ε, παλιότερα αναφέρει το χρονικό διάστημα τριών με πέντε ετών. Επίσης προτείνω οι επιτροπές αποδοχών να είναι εσωτερικές και ανεξάρτητες. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητες διότι εάν δεν είναι τότε ε, διότι αλλιώς μπορεί να λαμβάνει κανείς να διακινδυνεύει πολλά ε, σε περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητο. Ε, ξέρουμε ότι οι εισηγμένες εταιρείε ε, έχουν δυσανάλογα και πρόθεσμα μοντέλα αποδοχών, τα οποία τελικά οδηγούν στο να χάσει κόσμος τις δουλειές του, οι καταθέτες να χάσουν τις επενδύσεις τους ε, και οι επενδυτές ε, να πρέπει ε, να, επενδύσουν και άλλα χρήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε παρόμοια κρίση στο μέλλον και προσβλέπω στην καλή συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας και πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι όλοι ε, συμφωνούν με όσα προτείνεται. Ε, ε, σίγουρα μπορεί κάποιος να θέλει να υποβάλει τροπολογίες αργότερα, αλλά από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες παρατηρήσεις. 6 Μαΐου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 6 Μαΐου, σημαντική ημερομηνία, διότι ε, μπορεί κάποιοι από εσά να γνωρίζετε ότι έχουμε εκλογέ ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη μέρα. Τις ε, τροπολογίες θα τι εξετάσουμε την 1η Ιουνίου. Ε, θα το ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης την 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία στην ε, αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή ε, Οικονομικών ε, Υποθέσεων και προβλέπεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Κλείνουμε λοιπόν το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης και φτάνουμε στο ψήφισμά μου για την μακροχρόνια περίθαλψη. Πρόκειται για πρωτοβουλία που πήρα πριν αρκετό καιρό για διάφορους λόγους. Βασικά όμως επειδή πιστεύω ότι η μακροχρόνια περίθαλψη θα πρέπει να λάβει πιο σημαντική θέση στην ε, πολιτική ατζέντα. Όπως ξέρετε, η ε, κοινωνία μας γυράσκει και θα πρέπει να εξετάσουμε τους, τις συγκεκριμένες προκλήσεις ε, και τα θέματα που απορρέουν από το θέμα αυτό. Έχουμε την έκθεση του Τόμας Μαν, την οποία θα συζητήσουμε πρόσφατα. Έχω συνεργαστεί μαζί του ε, πάνω σε διάφορα από τα θέματα αυτά. Όσον αφορά την ε, συγκεκριμένη ερώτηση, παράγραφο 1. Ρωτώ την Επιτροπή τι ρόλο μπορεί να παίξει για τον καθορισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Πάντα θεωρούσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να κάνει περισσότερα όσον αφορά τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Στην παράγραφο 2 ρωτώ τι μπορεί να μας δώσει η Κομισιόν, τι στοιχεία μπορεί να μας παράσχει η Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των θανάτων ηλικιωμένων σε καθεστώς περίθαλψης, διότι φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων που πεθαίνουν από υποσυτισμό ή αφυδάτωση. Θα ήθελα πολύ να εξετάσω τα στοιχεία αυτά χώρα προς χώρα. Ξέρω αν είναι δυνατόν. Ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε Πολλού θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν και οι οποίοι αποδίδονται στον υποσυτισμό ή αφιδάτωση. Κάποιοι από τους ε, θανάτους αυτούς ε, τους έχουμε σε νοσοκομεία, άλλου, σε κέντρα περίθαλψης και άλλου, στα σπίτια ε, των ανθρώπων. Επίσης έχουμε τις εντολές μη ανάνυψης. Βλέπουμε αυξανόμενη χρήση των εντολών αυτών εντός της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και Κατά τη γνώμη μου, στην παρηγορητική γιατρική αυτό δεν είναι πρόβλημα και συχνά από εκεί προέρχονται. Αλλά όταν κάποιος ε, έχει λάβει διάγνωση για ε, μια ε, ασθένεια που θα οδηγήσει σε θάνατο, αυτό φυσικά είναι διαφορετική περίπτωση, διότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος και οι εντολές μη ανάνυψη στις περιπτώσεις αυτές είναι λογικές. Αλλά αν χρησιμοποιούνται σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ε, έχω πολλούς φόβους για το θέμα αυτό. Οι εντολές μη ανάνυψης δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ε, επιθυμία των ίδιων των ανθρώπων. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες οι εντολές μη ανάνυψης ε, δεν μπορούν να συμφωνηθούν από τους συγγενείς, από στο νόμο, σύμφωνα με τον νόμο δεν γίνεται αυτό και ο γιατρός θα πρέπει να τις ε, υπογράψει. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως οι συγγενεί έχουν ε, υπερβολικές ε, αρμοδιότητες όσον αφορά τι εντολές μη ανάνυψης. Αυτό λοιπόν είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε ε, λαμβάνοντα υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό είναι επίση ένα θέμα που θα πρέπει να θέσουμε πιο ψηλά στην ε, ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να σε αντικείμενο πολιτική συζήτηση, διότι δεν το συζητάμε αρκετά. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, οικονομικοί περιορισμοί σε πολλά κράτη-μέλη. Φοβούμε ότι τα νοσοκομεία και τα, ε, και τα γυροκομεία Ε, συχνά δεν παρέχουν ε, αρκετά ε, καλό βιωτικό επίπεδο και γι' αυτό θεωρείται ότι καλύτερα να μην συνεχίσει κανεί τη ζωή του. Θα ήθελα πάντως να συζητηθεί το θέμα των εντολών μη Ε, Στην παράγραφο 4 μιλώ για την κακοποίηση των ηλικιωμένων και ρωτάτε την Επιτροπή τι δουλειά έχει γίνει στον τομέα αυτόν. Ξέρω ότι έχει γίνει δουλειά στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη. Θα ήθελα Όμω πολύ να δω παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ε, κάποιων χωρών να εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε ε, τίποτα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την πρόληψη τη κακοποίηση ηλικιωμένων, είτε αυτή πραγματοποιείται στο σπίτι των ανθρώπων, είτε στον τομέα τη περίθαλψη, είτε στα νοσοκομεία. Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να λάβει πολλέ μορφέ, μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική ή οικονομική. Παράγραφος 5. Ζητά, ζητώ τη γνώμη της Επιτροπής ε, σχετικά με κώδικα συμπεριφοράς που να ε, ε, δίδει κάποιες ελάχιστες κατευθυντήρες γραμμέ και τα αποτελέσματα υπηρεσιών παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης. Αυτά όσον αφορά την προφορική ερώτηση. Ε, να προχωρήσω στην πρόταση ψηφίσματος ε, που για διαδικαστικού λόγου δεν μπορούσε να αποτελέσει το ίδιο σημείο στην ημερήσια διάταξη αλλά που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί. Στην παράγραφο 2 ε, αναφέρω ότι μαθαίνω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλα κράτη-μέλη αναφέρω Τονίζω το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή από εκεί προέρχονται οι μου εμπειρίες. Βλέπω ότι υπάρχει Περιορισμό στην ε, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και ε, καθώ επίση τη κατάρτιση των γιατρών ε, για, ζητήματα που αφορούν του ηλικιωμένου. Πολύ συχνά λέμε στου ηλικιωμένου ότι δεν είναι άρρωστο, απλά γερνάς. Και δεν λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα θέματα διάκριση των ηλικιωμένων ε, η γεροντική άνοια, το Alzheimer ε, είναι ε, ένα θέμα διότι συχνά η γεροντική άνοια δεν διαγιγνώσκεται. Απλά λένε στους συγγενείς ότι ο άνθρωπος γερνάει. Υπάρχουν όμως ε, θεραπείες ε, για την γεροτική άνοια και εάν ε, ξεκινήσει η περίθεση αρκετά νωρί, αν ξεκινήσει η θεραπεία αρκετά νωρί, τότε μπορεί να καθυστερήσει η εμφάνιση της νόσου. Θα ήθελα λοιπόν και εδώ να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από διάφορα κράτη-μέλη όπου δίδεται θεραπεία για τις περιπτώσεις αυτές, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν δίδεται. Ε, επίσης ζητώ εκτενέστερη έρευνα από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει υποσχεθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ε, τώρα πια μιλάνε για ε, διάσκεψη για την κακοποίηση ηλικιωμένων. Εγώ όμως θα ήθελα να δω πράσινη βίβλο, διότι έχοντα συνομιλήσει με συναδέλφους από ε, τα διάφορα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι κάτι που γίνεται γενικά, όπω σα είπα, και ε, σε σχέση με την προφορική μου ερώτηση. Η παράγραφος 5 ζητά καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω πάλι της ανοιχτής ε, μεθόδου συντονισμού. Όλοι ξέρουμε ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού αποτελεί... δεν ήταν τόσο επιτυχής όσο θα έπρεπε. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε στον κοινωνικό τομέα. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση σε άλλου τομεί, αλλά στον κοινωνικό τομέα πιστεύω ότι είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτήν, να την ενισχύσουμε και να την κάνουμε να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Μόνο όμως εάν έχουμε τη βούληση. Διότι όπως σας είπα υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που δεν έχει νόημα να ζητάμε νέα νομοθεσία στους τομείς αυτούς, ε, να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλον και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες αυτές τις πρακτικές. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, η μακροχρόνια περίθαλψη για τους ηλικιωμένους θα είναι οι υπηρεσίες στα όπως ε, και η παροχή υπηρεσιών υγείας που ε, έχουν ε, να κάνουν με ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιηθεί σε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την κοινωνία. Γι' αυτό ήθελα να θέσω το θέμα αυτό πιο ψηλά στην ημερησία διάταξη και ελπίζω μέσα στην επόμενη πενταετία να μπορέσουμε να εκπονήσουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς για όλα τα κράτη-μέλη για όλα τα θέματα αυτά που αφορούν τη μακροχρόνια περίθαλψη. Ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε οι ηλικιωμένοι στο τέλος της ζωής τους να μην αποκλείονται, να μην περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Φιγερέιδο και κατόπιν η Τζιν Λάμπερτ. Ε, κυρία αυτό το θέμα σχετίζεται το σημαντικό θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας. Γιατί για τους ε, ηλικιωμένους, στους ηλικιωμένους έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας επειδή λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, δεν έχουν συντάξει συχνά οι αποδοχές τους είναι υπερβολικά χαμηλές και γι αυτό, ήταν υπερβολικά χαμηλές και αυτό έχουν χαμηλή σύνταξη και ε, επίση τα προβλήματα των ε, γυναικών που είναι συνήθως τα πρώτα θύματα τέτοιου είδου ε, προβλημάτων. Οι γυναίκες ζουν και περισσότερο και αυτό δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα θετικό και δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα ε, και το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο, το συμπέρασμα μάλλον δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις κοινωνικές ε, παροχές αλλά και οι υπηρεσίε για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, οι κοινωνικέ υπηρεσίε για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά. Τόσο για του ηλικιωμένου όσο και για τα παιδιά. Γιατί και στα παιδιά έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό φτώχεια. Και αυτό δεν είναι απλή σύμπτωση. Εδώ χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα και το φαινόμενο αυτό χρήζει μια ιδιαίτερη προσοχή. Όπως είπαμε, οι αποδοχές είναι χαμηλές και σε πολλές χώρες η δημόσια υγεία καθώς και οι κοινωνικές παροχές δεν επαρκούν. Έτσι λοιπόν ε, καταλήγουμε σε φαινόμενα που περιέγραψε η Λίνα είναι σημαντικό να έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Είπα προηγουμένως ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την ε, παρούσα, την τωρινή κατάσταση των φτωχών. Η κοινωνική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά και τα παιδιά καθώς και ηλικιωμένοι πάσχουν ιδιαίτερα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κατεπηγόντως μια ενημέρωση των δεδομένων μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό τμήμα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Και εδώ δεν πρόκειται για μια σχετική ένδια. Σε πολλές περιπτώσεις πράγματι οι ηλικιωμένοι δεν, είναι, δεν βρίσκονται σε μια σχετική ένδια αλλά απόλυτοι. Και όπως σας είπα, όλα αυτά οδηγούν το να μην θέλει κανείς ε, να ζήσει εντολές μη ανάμνηψης, όπως είπε ο Μιλήτρη, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερο δαπανηρό για τα νοσοκομεία, για την υγεία κάτι που βεβαίω είναι ανεπίτρεπτο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη κατανομή του πλούτου. Και αυτά είναι πράγματι τα αποτελέσματα εσφαλμένων πολιτικών. Γι' αυτό είμαι απολύτως σύμφωνη με αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ. Γιατί πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί και μια παρόμοια πρωτοβουλία για τα παιδιά. Τα στοιχεία που μας ε, αναφέρατε πριν δείχνουν σε ποιο σημείο είναι η φτώχεια για των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προφορική ερώτηση υπάρχει ήδη ως πρόταση για να συζητηθεί στην ε, συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Να κάνουμε ακριβώς μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για τα παιδιά με στοιχεία σχετικά με αυτά που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, όπως ε, και για τους ηλικιωμένου που χρειάζονται ειδική βοήθεια. Και γι' αυτό ακριβώς και υποστηρίζω την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ. Εμείς καλωσορίζουμε την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Νομίζω ότι σε σχέση με τα όσα είπε μόλις η κυρία Φιγκερέντο, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι απαραίτητο υπάρχει σύνδεση με τη ένδια, αν και φυσικά έχει ρόλο να παίξει την ποιότητα της ζωής, όμως ε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η κοινωνική στάση, η κοινωνική συμπεριφορά. Πράγμα που αναφέρεται στην εισαγωγή της και γι' αυτό και πιστεύω πως η αναφορά στην προτινόμενη οδηγία για την ίση μεταχείριση είναι σημαντική, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο για... που αφορά τις διακρίσεις. Επίσης αφορά το θέμα της απομόνωσης. Δηλαδή, αν ε, κάποιος ε, μείνει μόνος του σε μια κατάσταση που κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία του, πραγματικά καθίσταται πολύ ε, ευάλωτος. Δεν θα καταθέσουμε πολλές τροπολογίες, αλλά μία μπορεί να αφορά την κοινωνική ένταξη. Και ίσως αυτή η διάσταση της κοινωνικής ένταξης θα ταιριάζει καλύτερα με την μέθοδο του συντονισμού. Επίσης θα ήθελα να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί παρακολούθησης Δηλαδή οι ηλικιωμένοι άνθρωποι όταν, αν είναι σε ε, γυροκομεία ή αν είναι στα σπίτια τους ε, πώς γίνεται η παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων ώστε να μην βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση όπου υπάρχει ατιμορρησία. Δηλαδή, κανένας δεν πρόκειται να έρθει να σε ψάξει ή να σε ελέγξει για μερικού μήνε. Και έχω και μια ερώτηση για το σημείο 1, όταν μιλάμε για την ειδική κατάρτιση για του επαγγελματίε και κατά πόσο αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης την ε, ε, βοήθεια και τη φροντίδα. Γιατί παλιότερα το έχουμε ξανασυζητήσει ότι θέλαμε να βελτιώσουμε την κατάρτιση και την κοινωνική θέση, το κοινωνικό κύρος αυτού του εργαζόμενου που φροντίζει για του γυραιότερου. Γιατί και αυτό είναι κομμάτι της, ε, των διακρίσεων. Θεωρείται γενικά μια δουλειά που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα και άρα δεν ε, του δίνεται σε αυτήν το βάρος που της αξίζει. Νομίζω λοιπόν πως είναι αυτή μια σημαντική πρωτοβουλία και το άλλο σημείο που ανέφερε η κυρία Φιγερέντο όσον αφορά τους νέους ίσως θα πρέπει αυτό το στοιχείο να το εντάξουμε σε κάποια μεταγενέστερη φάση. Ευχαριστώ η κυρία Γκόντσεφ. Σα ευχαριστώ και εγώ θέλω να καλωσορίσω την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό για μας που η κυρία Λίν έχει εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα ε, εδώ και πολλά χρόνια. Συμφωνώ και με το ψήφισμα και με την προφορική ερώτηση. Έχω απλώ μια ερώτηση. Μήπω θα ήταν σκόπιμο να τοποθετηθεί σε μια ευρύτερη κλίμακα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο σε σχέση με την ένδια που εσείς αναφέρατε, αλλά και σε σχέση με την ε, φροντίδα, την κοινοτική, ε, ούτως ώστε οι πιο ηλικιωμένοι να προτιμούν να μένουν σπίτια τους, να είναι μέρη δηλαδή της κοινότητας, από τη στιγμή που έχουν αυτή την υπηρεσία που τους ε, διευκολύνει να παραμείνουν. Και έπειτα εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για μέρημνα, για φροντίδα, να υπάρχουν ε, τα γυροκομεία ή οι ειδικέ ε, υπηρεσίες. Αυτό είναι μια πρόταση που θέλω να κάνω. Και έπειτα, το 2011 θα είναι το έτος ε, της ενεργής γύρανσης και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών. Από όσο γνωρίζω, και από τις πληροφορίες που έχω λάβει υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει. Είναι ένα άλλο ευρύ πλαίσιο και θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας να συζητήσουμε τα θέματα αυτά πιο εις βάθος, γιατί η... το ενεργό γύρας είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθήσει ακριβώς την ανάγκη για περαιτέρω φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Πρόκειται για τα στάνταρ της ε, μακροπρόθεσμης ε, φροντίδας ε, και πώς μπορούμε αυτό να τα λύσουμε. Θα ήταν ωστόσο χρήσιμο να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις πτυχές, αν συμφωνείτε. Πέρα από τον κώδικα διοντολογίας, ήθελα επίσης να αναφέρω τα minimum, τις μίνιμουμ προδιαγραφές ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που για το ποιος μπορεί να έχει τέτοιου είδους οίκους ευγυρία για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε αυτά να, τα, να θεσπίσουμε κάποιες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος θα σας απαντήσω. Κυρία Φιγερέδο, έχετε δίκιο. Μιλάμε για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και η Τζίν έχει δίκιο και αυτή σε, κατά κάποιο τρόπο ότι δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με την ένδυα αυτή καθ' αυτή αλλά σχετίζεται όπως εσείς είπατε με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί ποιες υπηρεσίες θα υποστούν περικοπές στα κράτη-μέλη. Θα είναι οι υπηρεσίες για τους ε, ηλικιωμένους και η μακροπρόθεσμη φροντίδα, η μακροχρόνια μάλλον ε, φροντίδα. σε, σε, οίκους Αλλά και στα σπίτια των ανθρώπων. Δηλαδή δεν λέω απαραίτητο πως θα είναι και ένα πλαίσιο οίκου ευγυρία, γυροκομείου ή νοσοκομείου. Γιατί έχετε δίκιο ότι αν κάποιος μπορεί να μείνει στο σπίτι του με κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος βέβαια. Από τη στιγμή που υπάρχουν όμως τέτοιου είδους υπηρεσίες. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια οικονομικά προβλήματα για τα κράτη-μέλη, πολλές φορές αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνο τους και άμεσα τοποθετούνται σε οίκους ευγυρία είτε στο νοσοκομείο. Και έπειτα ε, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για την λογοχώρα γιατί χρειάζεται να προσφέρει περισσότερη φροντίδα μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο. Αλλά έχουμε και την έκθεση που θα ασχοληθεί συγκεκριμένα με τις δημογραφικές αλλαγές. Θα μας απασχολήσει σύντομα. Για την οποία είναι ο Τόμας Μάνης ηγετής. Και στην έκθεση αυτή θα δούμε πολλά από αυτά τα θέματα. Νομίζω κάπου τον ε, Σεπτέμβριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Και επειδή φέτος έχουμε αυτό το χρόνο και προσπαθούμε να τονίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, είναι μια προσέγγιση βήμα προς βήμα. Εδώ έχουμε την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα και το Σεπτέμβριο θα έχουμε την έκθεση περί δημογραφικών προκλήσεων. Να μείνει δηλαδή το θέμα όσο γίνεται πιο πολύ καιρό στην ημερήσια διάταξη για την, την εκπαίδευση των ειδικών, των, των επαγγελματιών. Τους επαγγελματίες τους ε, ένταξε εδώ Εγώ σκόπευα να είναι όλοι μέσα εκεί, μαζί με τους, ε, τους ε, όλα τα επαγγέλματα φροντίδας ε, για τους ηλικιωμένου και μάλιστα αυτοί είναι που ασχολούνται με τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Ξέρω πως η, η κατάρτιση είναι όλα είναι και πιο υποβαθμισμένοι στα κράτη-μέλη για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δηλαδή κανείς δεν μπορεί να βρει δουλειά ως ταμεία στο σούπερ μάρκετ, βρίσκει δουλειά ως ε, ε, φροντιστής ηλικιωμένων. Και αυτοί που εργάζονται ε, αντίθετα σε αυτά τα επαγγέλματα ε, είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι. Επιλέγουν να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί θέλουν να τη κάνουν συνήθως και νομίζω πως θα πρέπει να αναγνωριστούν και όχι μόνο να αναγνωριστούν αλλά να έχουν και στις δικές τους προδιαγραφές κατάρτισης και αν μπορούσαμε να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες ευχαρίστως θα το κάνω να πούμε δηλαδή ότι αυτού του είδους η δουλειά θα πρέπει να αναγνωριστεί όπως της αξίζει και όχι να λένε ή και ευγυρίε ότι ναι, χρειαζόμαστε περισσότερου φροντιστέ, αλλά δεν, επειδή δεν του έχουμε. Αλλά δεν τους έχουν γιατί ακριβώς δεν τους πληρώνουν τα κατάλληλα, τους κατάλληλους μισθούς και δεν ε, ε, τηρούν τις κατάλληλες ε, συνθήκες. Ξέρω, σε πολλούς οίκους ευγυρίες, ακόμα και αν δουλεύουν υπερορίες, πρέπει να πληρώνουν για το φαγητό τους. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή το γυροκομείο να, έχει, να ετοιμάζει φαγητό για τους οικότροφους και για το προσωπικό και ιδιαίτερα για τους φροντιστές, τους νοσοκόμους. Οι νοσοκόμοι μπορεί να παίρνουν το φαγητό, να τους δίνουν, τους προσφέρει το φαγητό τους, αλλά οι, δική βοηθοί αυτοί οι φροντιστές άντε να πάρουν κανένα σάντουιτς και πολλές φορές και τίποτα. Θυμηθείτε πως πολύ συχνά παίρνουν την, την, τους ελάχιστους μισθούς. σε πολλά Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε όχι μόνο να πάει καλά η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα, αλλά όταν θα πάρουμε την έκθεση για τις δημογραφικές αλλαγές, προκλήσεις, να μην το αφήσουμε αυτό εκτός της εξίσωσης. Ξέρω ότι ο τόμα Μαν λοιπόν κοιτάει το θέμα, εξετάζει αυτό το θέμα και όλε οι παρατηρήσει που κάνατε είναι πολύ σημαντικέ νομίζω. Ευχαριστώ. θα συνεργαστώ μαζί σας για τροπολογίες γιατί είναι πολύ σημαντικό το αρχικό στάδιο να το φτιάξουμε σωστά και να προχωρήσουμε με τον Τόμας και να δουλέψουμε για τα ευρύτερα ζητήματα για, στην έκθεση για τις δημογραφικές προκλήσεις. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαστε μισή ώρα μπροστά. Οι ψηφοφορίες είναι στις 11. Νομίζω λοιπόν πως είναι καλή ιδέα να κάνουμε ένα μισάωρο διάλειμμα, να είμαστε πίσω στις 11 ακριβώς για τις ψηφοφορίες. όσο μόνο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 Παρακαλώ καθίστε όλοι. Πριν από την έναρξη των ψηφοφοριών θα ήθελα να σας ζητήσω να, προχωρήσουμε, να κάνουμε μια δοκιμή ώστε να επαληθεύσουμε πως όλοι έχουν τις κάρτες τους και ότι κάθε πολιτική ομάδα έχει τους ε, βουλευτές της εδώ αλλά χωρίς να έχει παραπανήσιους. Τώρα το ποιος θα ψηφίσει αυτό μεταξύ σας θα βρείτε τα.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 έχω την αμυδρά εντύπωση ότι ψηφίσαν περισσότεροι από όσοι μπορούν να ψηφίζουν. Oui, mais sauf que dans le pas une petite attaque. Donc, alors, euh, je clôt le vote. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Και είχαμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω και έξι ΕΛΚ. Έξι. Donc, Φαντάζομαι ότι λοιπόν ανάμεσα στους ε, ε, αναπληρωματικούς του έλκα πρέπει λίγο να τα βρείτε. Λοιπόν, για βάλτε τάξη εκεί στο ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές το ίδιο είναι πιο εύκολο γιατί είναι ένας μόνο. Bien. Est ce que je peux demander au coordinateur du groupe PPE si nous pouvons reprendre nos... Να ρωτήσω το συντονιστή του ΕΛΚΑ αν μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Maintenant, je crois qu'il nous να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Αν θέλει να καθίσει και ο κύριος Ορή, θα κάνουμε μια νέα Παρακαλώ. Ψηφίζουμε. τέλος ουφορίας βλέπω δύο έλκα παραπάνω. Έρχεται και η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Κύριε Ορή, παρακαλώ βιαστείτε. Βάλτε τάξη εκεί στις ε, γραμμές σας. Να μην... Να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 Δεν θέλω εγώ να μπω τώρα να βάλω τάξη στο ΕΛΚΑ, ε, οπότε ε, ας κάνουμε μια τελευταία δοκιμή. Tout Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Ωραία, τα καταφέραμε. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτη έκθεση από της οποίας πρέπει να ψηφίσουμε είναι έκθεση της κυρίας Έντιτ Μπάουερ για την οργάνωση του χρόνου εργασία. 16, 17 και 18 είναι οι, προτα... οι προτάσεις απόρρεψης της ε, ε, έκθεσης. Το ψηφίζουμε από κοινού. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 49 ψήφισαν, 30 υπέρ, 19 κατά. Le rapport de Madame Edith Bauer est rejeté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 Μείνετε στις θέσεις σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε την απόρριψη της πρότασης, ψηφίσαμε μάλλον την πρόταση απόρριψης της, προ, της ε, πρότασης της Κομισιόν και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε και για το ίδιο το νομοθετικό ψήφισμα. Είναι στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας σας. Ψηφίζουμε λοιπόν. την νομοθετική πρόταση όπως τοποποιήθηκε. Όσοι είναι υπέρ της πρότασης απόρρευσης ε, της Κομισιόν θα πρέπει να... Κυρία Χάρκιν. το συγγνώμη, Πρόεδρε αλλά δεν κατάλαβα ακριβώ τι ε, ψηφίζουμε. Ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Αν και είμαστε στα μέση μιας ψηφοφορία. και δεν θα έπρεπε να τη διακόπτουμε. Λοιπόν, ψηφίσαμε την απόρριψη της νομοθετικής πρότασης. Όχι, ψηφίσαμε την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε με τελική ψήφο για την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος στο σύνολό της. Πράγμα που σημαίνει ότι όσοι είναι κατά τις θέσεις της κυρίας Μπάουερ πρέπει να καταψηφίσουν. Bien. Alors, on va... Excusez-moi. Il y a eu une toute petite confusion et on va essayer de Συγγνώμη, υπάρχει μια επικρατή μια σύγχυση. Αν δείτε το κατάλογο ψηφοφορία σα, μετά από την εξέταση του συνόλου των τροπολογιών στην έκθεση τη κυρία Μπάουερ, έπρεπε να καταλήξουμε σε μια τελική ψηφοφορία για το σύνολο τη έκθεση τη κυρία Μπάουερ. Η έκθεση τη κυρία Μπάουερ τώρα συμπεριλαμβάνει μόνο ένα άρθρο, δηλαδή την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν. Να. Σας προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Μπάουερ καθ... όπως τροποποιήθηκε. Λοιπόν, συμφωνείτε. Le vote est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter? Ψηφίσατε όλοι. Le vote est clos. Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 19 κατά, καμιά αποχή. Nous en venons au dernier vote. Τελευταία ψηφοφορία που είναι τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα το νομοθετικό. Όπως το Même, même, même motif, même punition. C'est-à-dire que Όσοι είναι υπέρ της απόρριψης πρέπει να ψηφίσουν υπέρ. Tout le monde a pu voter, le vote est Ψηφίσατε όλοι, τέλος Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Και έτσι τελειώσαμε με αυτή την ψηφοφορία. Και τώρα έχουμε τη γνωμοδότηση του συναδέλφου Χάουιτ για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα κοινωνικά και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Έχουμε την τροπολογία του κ. Κάσλερ, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική α, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3 του κ. Higgins, που είναι συμβατή, υπέρ, κατά, αποχές, Επαληθεύουμε. Τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. 19 ε, υπέρ, 26 κατά. Παράγραφος 2, τροπολογία 5. Κάσλερ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 ρίνιε υπέρ κατά νομίζω πως εγκρίνεται. 5 Higgins. Να το επαληθεύσουμε, εντάξει, αφού θέλετε να το επαληθεύσουμε για την 6. Τέλος ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Higgins, 7. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, δεν είναι σαφές. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8, του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Αποχές, νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 8. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οι 9 και 11 είναι συμβατές. Καταρχήν η 9 της κυρίας Ράπτη, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 της κυρίας Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 12 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. παράγραφο euh, Τροπολογία 16 και 15 είναι για διαγραφή. Υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική Β, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 14 πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, ε, ψηφίζουμε για τη 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6. Παράγραφος 6. Τροπολογία 19. Χίγγινς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. κάστλερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, ήταν το 20. Όταν το καταλάβω ήταν το 20. Λοιπόν, στην παράγραφο 6, τροπολογία 20 Κάστλερ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική σε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, συμβιβαστική, D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική D εγκρίνεται. Παράγραφος 8, 20, 25 του υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 25 ηλεκτρονικά. Τέλος πληροφορίας, 27 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν για ένα τμήμα της 26 που δεν καλύπτεται από την 25 που λέει με εμπλοκή των αντιπροσωπών των εργαζομένων και των κοινωτικών οργανώσεων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27, 9 είναι συμβατή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 9, την τροπολογία 29, Κάστλερ, για διαγραφή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 32, Κάσλερ, περ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Τροπολογία 32. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Καταπίπτει η 32. Και έκανα λάθος, σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Έπρεπε να ψηφίσουμε και για την τροπολογία 31 που δεν έχει καταπέσει. Λοιπόν την ψηφίζουμε. Την 31 για την παράγραφο 9 ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Τροπολογία 32 δεν έχει εγκριθεί. Οπότε ψηφίζουμε για 33 του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας. Έχουμε τη 34 τώρα του κυρίου Τόμας Μαν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 24 υπέρ. 21 κατά, 3 αποχές να συγχαρούμε τον εισηγητή μας. περάσουμε στη ψηφοφορία για την γνωμοδότηση για την έκθεση, συγγνώμη, λέει ομιλία, ομιλήτρια, του κυρίου, η πρόεδρος του κυρίου Σέρκας. Ε, το εννέο αίτημα για χορήγηση άδεια εργασία και διαμονή. Άρθρο 2 Β. Τροπολογία υπαριθμών 24. Δύο συντάκτε. Τροπολογία 24 χωρίς το στο πλαίσιο μιας αμοιβόμενης σχέσης. που θεωρείται ασύμβατες με το πεδίο αρμοδιότητας της, Επιτροπή της Επιτροπής μας ε, και την άποψη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Λοιπόν, υποβάλλεται σε ψηφοφορία χωρίς αυτή τη διατύπωση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Σιγητά, Κυρία Πρόεδρε, ήθελα απλώς να σας πω, γιατί μου το ζήτησε ο Τόμας Μαν, να διευκρινίσω ότι οι συμβιβασμοί που θα ψηφίσουμε σήμερα περιλαμβάνονται στην τροπολογία 25 του Τόμας Μαν μέχρι την τελευταία παράγραφο. παράγραφο. Είναι ένα συμβιβασμό όχι για την αιτιολογική σκέψη 12 μόνον, αλλά και για την τροπολογία 25 του Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση. Υποβάλλουμε λοιπόν σε ψηφοφορία το συμβασμό Α που αφορά το 12 και την τροπολογία 25 του Τόμας Μαν. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, παράγραφος 1, Σημείο 1, 26 του Λαϊαρή και άλλων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Ε, ψηφίσατε άπαντες, ωραία. Λύεται ψηφοφορία. 49 υπέρ, εγκρίνεται. η κυρίας Γκρουνή, 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 του εισηγητού. Όχι, κατά 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα κάνουμε επαλήθευση, τροπολογία του εισηγητού. Νομίζω ότι είναι η ίδια ψηφία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία παριθμών 6. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 20 υπέρ υπέρ, 28 κατά, έχετε δίκιο, δεν εγκρίνεται. 28 της κυρίας Όιμαν Ρόικεν, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 29 καταπίπτει. Οκτώ του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 της κυρίας Μάισνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 του εισηγητού καταπίπτει 31 του Τόμας Μαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 της κυρίας Τζιν Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επαλήθευση για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 28 κατά. Απορρίπτεται. Η 32. Ναι, επί του κανονισμού, επί διαδικαστικού θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κοιτάτε πραγματικά τα χέρια που υψώνονται. Γιατί όλο λέτε εγκρίνετε, απορρίπτεται αποχές χωρίς καν να ρίχνετε ένα βλέμμα στα χέρια. Και επειδή κάνετε λάθος δύο φορές, θα ήθελα να επιδείξετε μεγαλύτερη αυστηρότητα στην άσκηση του καθήκοντός σας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για αυτή την παρατήρηση, θα τη λάβω υπόψη μου. Τώρα, Περνάμε στη 10 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. του κυρίου Λεγιαρίκ και 34 της κυρίας Τζιν Λάμπερτ για διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχή, απορρίπτονται. 11 του εισηγητού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 του εισηγητού και 35 του κ. Λοϊαρίκ. Ε, τις υποβάλλω από κοινού σε ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχής, θα επαληθεύσουμε. Οι 35 και 12. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες, 21 ψήφοι υπέρ, 29 κατά. Δεν εγκρίνονται. 13 του εισηγητού και 36 του κυρίου Λοϊαρίκ και άλλων επίσης για διαγραφή. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία αλλά θα επαληθεύσουμε όταν ξεμπλοκαριστεί το σύστημα. Ωραία, λοιπόν, θα μπορέσουμε να κάνουμε την επαλήθευση 13 και 36. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 26 ψήφοι πέρα, 24 κατά και μία αποχή αλλά υπάρχει ένας ε, σοσιαλιστής παραπάνω. Δηλαδή 26 συν ε, υπέρ 23 κατά και μία εποχή. Οι τροπολογίες 13 και 26 εγκρίνονται. Donc le η συμβιβαστική τροπολογία καταπίπτει. Και θα πράσουμε στη ψηφοφορία για την 38 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές ε, επαλήθευση 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 40 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Η τροπολογία 38 εγκρίνεται. 14 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. στην αιτιολογική σκέψη 9, τροπολογία 16, στις ίδιες συνθήκες όπως και η προηγούμενη ψηφοφορία, χωρίς ε, το ε, στο πλαίσιο μιας αμοιβόμενης σχέσης. Ποιος είναι υπέρ της 16. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ένα του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 του Λεαϊαρίκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 της κυρίας Μπλίνκεβιτσιωτέ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 έχει καλυφθεί από τη συμβαστική τροπολογία Α. Θα περάσουμε λοιπόν στη τελογική σκέψη 16. Ε, τροπολογία Γ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καταπίπτουν και θα περάσουμε μετά την ιδεολογική σκέψη 16 στην τροπολογία περιθμών 22 που θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Καταρχήν το πρώτο τμήμα η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει μέχρι με τον ε, νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το υπόλοιπο τμήμα του κειμένου υπέρ. Υπέρ. Ε, ο εισηγητής είναι κατά. Για το δεύτερο τμήμα του κειμένου υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Κυρία Όιμεν Ρόιτερ, θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την 23 της κυρίας Τζιν Λάμπερτ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. κυρία Όιμεν Ρόιτερ, θέλετε να παρέμβετε. Ε, κυρία Πρόεδρε, ως ε, ΕΛΚ κάναμε ένα λάθος σε σχέση με τροπολογία υπαριθμών 13 με τον συνάδελφο κύριο Σέρκας και άλλους συναδέλφους ε, είπαμε ότι είμαστε κατά, γιατί εξ αρχής είμαστε, ε, αρχικά συγγνώμη, είμαστε κατά, αλλά στην διαπραγμάτευση για τους συμβιβασμούς είπαμε ότι θα το καταψηφίσουμε. στο κατάλογο ψηφοφορίας, ε, το κατάλογο ψηφοφορίας δυστυχώς δεν τον εξέτασα. Ε, λυπούμε νόμιζα ότι θα είναι σωστός. Αλλά εδώ για το 13 υπάρχει ένα συν, μια υπερψήφιση. Και τώρα η τροπολογία έχει υπερψηφιστεί, ούτως ώστε να διαγραφεί το κείμενο της Επιτροπής. Αλλά είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βρούμε εδώ μια λύση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να παρακαλέσω και τους συναδέλφους να αναβληθεί και ίσως να επαναληφθεί κάποια άλλη φορά. Euh, ναι, είναι μια έκτακτη κατάσταση. Στη γαλλική νομοθεσία υπάρχει ένα προνόμιο της ε, γαλλικής κυβέρνησης η οποία μπορεί να ζητήσει μια δεύτερη διαβούλευση. Σας προτείνω μια διαβούλευση λοιπόν των μελών της Επιτροπής για να επαληθεύσουμε κατά πόσο, αν υπάρχει ένσταση ή όχι, για να περάσουμε σε μια δεύτερη ψηφοφορία για την παράγραφο 13 και την τροπολογία 26. Στην περίπτωση αυτή θα ψηφίζαμε την παράγραφο Β. Δεν ξέρω, κύριε Σιγητά, θέλετε να μας ε, να φωτίσετε την κατάσταση. Ναι, κυρία Πρόεδρε με το ίδιο αποτέλεσμα, ίσως υπάρχει κάποιος άλλος ε, δρόμος πριν λογικός. Δηλαδή, να ψηφίσουμε πρώτα το συμβιβασμό και αν υπερψηφιστεί θα καταπέσουν οι τροπολογίες. Συμφωνούμε με την ε, διαδικασία του ΕΛΚ, το οποίο ε, έσφαλε. Κύριε Σιγητά, συμμερίζομαι πλήρως την άποψή σας εφόσον υπάρχει μια συμβιβαστική τροπολογία καταπίπτουν οι άλλες αλλά η αυστηρή ανάγνωση, η αυστηρή ερμηνεία δηλαδή όταν υπάρχει μια ε, τροπολογία που, απόρριψης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια συμβιβαστική τροπολογία αλλά όλα αυτά από μια ε, επιστήμη που δεν είναι η δική μας, τώρα που βρισκόμαστε εν μέσω μιας ψηφοφορία. Γι' αυτό κατανοώ τη θέση σας. Κυρία ε, Ρόιτερ, εφόσον ικανοποιώ το έτοιμά σας, δεν χρειάζεται να ξαναπάρετε το, ρόλο σας, ε, το λόγο. Θα ξαναψηφίσουμε την 13 και 36 και μετά την παράγραφο Β. 13 και 36 ψηφίζονται τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Ωραία, λοιπόν, τώρα εγκρίνεται από 8 και απορρίπτεται από 41, άρα απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στη συμβαστική ε, ε, ψηφοφορία, συμβαστική τροπολογία Β, στο συμβασμό Β. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 4 αποχέ, άρα ο συμβασμό Β εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Ρόιτερ για τη συμβολή σα σε αυτή τη συλλογική εργασία. Παρ' όλα αυτά θέλετε να έχετε το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά σας προσωπικά αλλά και τους συναδέλφους για την διάθεση να, που έδειξαν να συνεργαστούν εδώ. Αλλά το δεύτερο είναι το εξή. Δεν θα έπρεπε να ψηφίσουμε πρώτα για τη συμβαστική τροπολογία και μετά τις τροπολογίες. Αυτή ήταν η παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Κυρία Όιμαν Ρόιτερ, έθεσα αυτό το ζήτημα ε, αφορά το, θεωρία και θα ήθελα η γραμματεία να επαληθεύσει του πώς θα πρέπει να παρουσιάζονται οι τροπολογίες όταν υπάρχει μια τροπολογία κατάρριψης. Ε, απόρριψης. Συγγνώμη. Ε, θα πρέπει να μας πει η γραμματεία τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι νομικό το θέμα. Και συμφωνώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή μου κάνει εντύπωση το γεγονός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει επίτευξη ενός συμβιβασμού, είναι ισχυρότερος από την απόρριψη η οποία είχε οικοδομηθεί στη βάση της επίτευξης του συμβιβασμού. Αλλά εάν θέλετε μπορούμε να προσφύγουμε στις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επαληθεύσουμε αυτή την ερμηνεία του κανονισμού και το ορθόν της ψηφοφορίας. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Κύριε Σεγητά, ίσως έσφαλα αλλά νομίζω ότι δεν ψηφίσαμε την 23 ε, της ε, Jean Lambert. Όχι, ε, την ψηφίσαμε. Τώρα θα δώσουμε, θα περάσουμε στην οριστική ψηφοφορία που γίνεται ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, 42 ψήφοι υπέρ, μία αποχή, μία ψήφος κατά και επτά εποχές. Μπορούμε να σας συγχαρούμε κύριε Σέρκας. Βρισκόμαστε σε μια συνδεδεμένη διαδικασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως διατυπώνεται επισήμως. Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις δηλαδή με το Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε τον εισηγητή να συμμετάχει στη διαπραγμάτευση στη βάση αυτής της ε, τελικής γνωμοδότησης έτσι όπως μόλις την εγκρίναμε. Έτσι λοιπόν οι δύο αυτές δυνάμεις μπορούν να ενωθούν για την διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Η ψηφοφορία για το σημείο 18 έχει αναβληθεί, έτσι όπως είπαμε χθες, και θα περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Τσίμερ για τη μείωση της ε, φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση την οποία Ε, συντάξαμε υποβάλλουμε στην Επιτροπή ε, Ανάπτυξης. Παράγραφος 1, τροπολογία 1 της κυρίας Ντέλη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 της Ιδίας, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 της κυρίας Ζίπελ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 της κυρίας Ντέλη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 της κυρίας Τσίμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 της ιδείας υπέρ κατά εγκρίνεται 7 της κυρίας Τσίμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 της κυρίας Ζήπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 της κυρίας Γιαρόκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, της κυρίας Τσίμερ 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 11 της κυρίας Τσίμερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 12 της κυρίας Γκρινή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 13 της κυρίας Γιάροκα υπέρ, κατά αποχές, έχω την εντύπωση ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε παλήθευση. Για την 13 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι πέραση τη ψηφοφορία. 24 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Η τροπολογία υπαρθμών 13 εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην τροπολογία υπαρθμών 14 της κυρίας Ζίπελ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 της ιδείας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 7 τοπολογία 18 της ιδείας υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 έως 27 μπορούν να ψηφιστούν από κοινού όχι ωραία 20 της ηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 της ηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 της ιδίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 23 της κυρίας Τσίμερ. «23». Να επιβραδύνω λοιπόν το ρυθμό. Ωραία. Θέλετε μια επαλήθευση για την 22. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 25 ψήφοι υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται, έστω και με κάποιους ε, ενδιασμούς. 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24, τη ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25, Τη εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επαλήθευση για 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στι ψηφοφορίες. 23 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται με μικρή πλειοψηφία. 26 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 43 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, μία εποχή. Νομίζω ότι μπορούμε να συγχαρούμε την εισηγήτριά μας. Bien. Euh, euh, Τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση. Το ψήφισμα για την κοινωνική διάσταση τη ε, στρατηγική 2020. Για την προφορική ερώτηση, καταρχήν, τροπολογία υπαριθμών 1 τη κυρία Λίν. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 2 τη κυρία Λίν. Υπέρ. Αποχέ εγκρίνεται. Το σύνολο τη προφορική ερώτηση υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην ψηφοφορία του ψηφίσματος παράγραφος 1, τροπολογία 6 του κυρίου Καπνόχ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κύριε Ρίβ, θέλετε επαλήθευση για το 6, για την 6. Επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας στις ψηφοφορίας. 17 ψήφοι υπέρ, 25 ψήφοι κατά, μία αποχή. Δεν εγκρίνεται αυτή η τροπολογία. Και τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 1 με μία προφορική τροπολογία που υπέβαλαν οι πράσινοι και το άλτε. Υπέρ αυτές της τροπολογίες της παραγράφου 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται μετά την παράγραφο 3 μια τροπολογία υπαριθμών 7 του κυρίου Καμπρινόχα. Σας προτείνω εδώ μια προφορική τροπολογία. Δεν έχετε καμία αντίρρηση. Ωραία, η 7 όπως έχει τροποποιηθεί υποβάλλει σε ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο, θα παρεθεύσουμε. Η 7 ως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορία 7 ψηφί πέρα 37 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά, ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 8 του κ. Καπρνόχ, υπέρ. Κατά, αποχέ. απορρίπτεται. Παράγραφο 4, τροπολογία 9, την κυρία ε, Σαν και όπου το, η διατύπωση ε, κύριος, main, θα αντικατασταθεί από το σημαντικό, an important. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 10 της των ιδίων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται μετά την παράγραφο 4, πάλι 11 των ιδίων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, παράγραφος 5, σημαντική τροπολογία α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία της κυρίας Μπιζότο σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Μέχρι την αριστεία των πρακτικών και των περιεχομένων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το υπόλοιπο τμήμα του κειμένου. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο για το 15 του κυρίου Καπρινόχ υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε για το 15. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 26 ψήφοι Πέρα 17 κατά. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 7 ε, τροπολογία 17 της κυρίας Λίν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 της κυρίας Χάρκιν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δε. Με την παράγραφο 7, τροπολογία 19 της κυρίας Κόρνελ Σεν και του Ρούνεν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, 20 τη κυρία Χάρκιν, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 9, συμβασική τροπολογία Β, πουρ. Ε, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 22 της κυρίας Κόνησεν και του Ρούν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, 25 της κυρίας Λίν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 15, αρπολογία 26 του κυρίου Καπνόχ. Υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την αρπολογία παριθμών 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφορίες. 23 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 4 αποχές. Η τροπολογία υπερθυμών 26 εγκρίνεται. 27 του κυρίου Κάρπνοχ υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται στην παράγραφο 16 η τροπολογία 28 της κυρίας Λίν υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 29 της κυρίας Αρκίν, είναι συμβατή υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 17 τροπολογία 30 της κυρίας Λίν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 τροπολογία 31 της κυρίας Λίν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 της κυρίας Αρκίν συμβατή υπέρ κατά θα παληθεύσουμε 32 Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας 26 ψήφοι 5 17 κατά εγκρίνεται μετά την παράγραφο 18 τροπολογία 33 των κυρίων Κόρνελσεν Ρούνεν σε δύο τμήματα. Πρώτα το πρώτο τμήμα, Καλή το Συμβούλιο κλπ. Invite the Καλεί το Συμβούλιο και λοιπά, συνδυάζοντας έργο και κατάρτιση. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα το δεύτερο τμήμα. Το υπόλοιπο της 53 υπέρ κατά αποχές επίσης συγκρίνεται μετά την παράγραφο 18 34 των ιδίων υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για 34 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας 20 ψήφοι υπέρ 24 κατά απορρίπτεται παράγραφος 19 35 γλυκά πνόχα για διαγραφή υπέρ κατά άπτεται 36 ρεαλίν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Για 37 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. όλοι ψηφοφορίας. 20 ψηφί 23 κατά. Απορρίπτεται. Τραπολογία 38 των ιδιών υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίζεται πλέον πολύ. Θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Η 39 του, των ιδίων υπέρ, κατά. Αποχές, η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. 40 του κυρίου Καπρινόχ υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 κυρίες Λίν υπέρ, ε, εγκρίνεται, 42 τη κ. Χάρκιν ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 των Κορνέλη Τουρίνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 24, τροπολογία 24 των Ινδίων υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε για τις 44. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 25 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 24, τροπολογία 45 τη κυρία Λίνη. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Τροπολογία για, καταστολή του κυρίου, ε, για διαγραφή του κυρίου Καμπρινόχα υπέρ τη 47 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26, 56 του κ. Καπρινόχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 της κ. Ζηλίνη. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 27 τροπολογία 51 του κ. Καπρινόχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 της κυρίας Λινιπέρ. Κατά κατά αποχές εγκρίνεται 52 της κυρίας Αρκίνη Πέρ. κατά αποχές εγκρίνεται πράξη 28 τροπολογία 53 των κυρίων Κορνέλησεν του Ρούναν υπέρ κατά αποχές θα παληθεύσουμε την 53 Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 18 ψήφοι υπέρ, 23 κατά. Η 53 δεν εγκρίνεται. 54 της Λίν υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται παράγραφος 29, τροπολογία 55 της κυρίας Μπιζότο. Με μια προφορική τροπολογία δική μου. Όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά αποχές Θα επαληθεύσουμε. Για την 55. Ψηφίσατε όλοι, Πέρα ψηφορίες, 40 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και 30 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, αιτιολογική σκέψη Β. κονέλησαν του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γ. Αιτιολογική σκέψη Γ. 2 του κ. Καπνόχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 την κυρία Κορνίλησεν του Ρούνεν μετά την λογική σκέψη γάμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 των ιδίων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 των ιδίων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Κύριε Ρή, έχετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα απλά να τονίσω μετά την ψηφοφορία ότι δεν συμφωνούσαμε να μπει αυτό στην ημερήσια διάταξη και δεν μας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα και γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής των Συντονιστών είναι υπέρ. Ε, νομίζω ότι είναι δεδειγμένο να συζητήσουμε εδώ τη στρατηγική 2020 στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής και πρόκειται να την υπερψηφίσουμε. Τίποτα άλλο, επεξηγήσεις ψήφου άλλε. Όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και ολοκληρώσαμε έτσι τις ψηφοφορίες μας. Σας ευχαριστώ και ραντεβού στις 3 για την εξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών για την έκθεση του κυρίου Όρη.